Very Καλή σας μέρα όλοι. Καλώς ήρθατε στην σημερινή μας ψηφοφορία. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτήν την δύσκολη μέρα. Πριν αρχίσουμε όμως τις ψηφοφορίες, θα ήθελα να είσαστε σίγουροι ότι έχετε μαζί σας τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Έτσι. Αυτή είναι η τελευταία συνεδρίαση μετά από ένα χρόνο εντατική δουλειά που έχουμε κάνει στην Επιτροπή μα. Ξεκινήσαμε με τη συγκρότησή μα σε σώμα στι 22 Μαρτίου, πριν από ένα χρόνο δηλαδή. Θέλω να σας υπενθυμίσω πόσο πολλή δουλειά έχει γίνει στην Επιτροπή μας. Ξέρετε ότι είχαμε 34 συνεδριάσεις 18 δημόσιες ακροάσεις, 10 ανταλλαγές απόψεων με εκπροσώπους των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των χωρών μελών, τρία εργαστήρια και τρεις συζητήσεις επίσης στα πλαίσια της ε, σύνταξης αυτής της έκθεσης. Συλλέξαμε, αναλύσαμε πάρα πολλά στοιχεία που λάβαμε και γραπτά και προφορικά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, όπως επίσης και από μελέτες που αναθέσαμε και βεβαίως και από τις τέσσερις αποστολές που πήγαμε, διαρευνητικές, που οργανώθηκαν από την Επιτροπή μας στη Ουάσιγκτον, στη Λετωνία, στο Isle of Man, στην Εστονία και τη Δανία. Πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι τα συμπεράσματά μας συμπεριλαμβάνονται στις συμβαστικές προτάσεις που θα ψηφίσουμε σήμερα. Θα ψηφίσουμε σήμερα κάτι που αντικατοπτρίζει πάρα πολύ καλά τις θέσεις της Επιτροπής μας μετά από τα θέματα τα οποία εξετάσαμε εδώ κατά τη διάρκεια της εντολής μας. Θέλω να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές, τον Λούντεκ Μάιερ και τον Γεπε Κοφόντ για το έργο τους. Πράγματι η εντολή της Επιτροπής μας αυτή ήταν εκτενή και καλύψαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Το σχέδιο έκθεσης κυκλοφόρησε στις 14 Νοεμβρίου που μας πέρασε. Η εξέταση, η συζήτηση του σχεδίου αυτού έκθεσης έγινε στις 27 Νοεμβρίου εδώ στην Επιτροπή μας του 2018. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ήταν 17 Δεκεμβρίου και η γραμματεία έλαβε σχεδόν 1.300 τροπολογίες. Η εξέταση των τροπολογιών έλαβε χώρα στη συνεδρία της Επιτροπής μας στις 29 Ιανουαρίου. Οι συνεισηγητές λοιπόν, βάσει αυτών, συναντήθηκαν πολλές φορές με τους σκιώδεις εισηγητές και πρότειναν τελικά 150 συμβαστικές τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης. Οι συμβαστικές αυτές προτάσεις έχουν μοιραστεί από τη Γραμματεία έγκαιρα. Θα δώσω το λόγο στους δύο συνεισηγητές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, ολοκληρώνουμε τώρα όχι μόνο το έργο της Επιτροπής Ταξ 3, αλλά και γενικώ το έργο μας στον τομέα της φορολογίας κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτέλεσε εξαιρετικό έργο και ενίσχυσε την γνώση μας όσον αφορά το θέμα και έτσι ε, μπορεί να σταθεί και μπροστά στους ε, πολίτες για έναν τομέα που είναι πάρα πολύ σημαντικός για την οικονομία και την πολιτική στην Ευρώπη. Όσο δουλεύαμε πάνω στην έκθεση αυτή, όπως ε, πολύ σωστά είπατε, προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Χρειάστηκε να συγκλίνουν οι απόψεις μας και να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει, όλες οι πολιτικές ομάδες δηλαδή. Όσοι συμμετείχαν, όντως έχουν πολύ καλές γνώσεις στο θέμα. Σίγουρα παραμένουν κάποιες διαφορές μεταξύ μας, όμως, διακόπτει ο Πρόεδρος, παρακαλώ ησυχία στην αίθουσα. Έλεγα λοιπόν ότι το βασικό μήνυμα και η σημασία του θέματος είναι κάτι τα, με, σχετικά με το οποίο συμφωνούμε όλες οι πολιτικές ομάδες εδώ στο Σώμα και αυτό ήδη είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν. Πρώτα απ' όλα τον συνεισηγητή μου, Ιαν Κοφότ και τους συνεργάτες του. Αλλά να πω επίσης ότι η συνεργασία μου με τους σκιώδεις ήταν εξαιρετική. Πέρασαν όλοι ώρες μαζί μου προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβασμούς και λύσεις. Αυτή δεν είναι μια έκθεση για το ΕΛΚ ή για του σοσιαλιστέ. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή έκθεση για την Ευρώπη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ επίση τη γραμματεία, των Μπενουά πρώτα απ' όλα και του ε, δικού του συνεργάτε για τη βοήθειά του. Επίση, ο Γιάννα Έριξ Μαρτίνα και η γραμματεία του ΕΛΚ, οι συνεργάτε μου δηλαδή από το ΕΛΚ, με βοήθησαν πάρα πολύ και του ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διέθεσαν στην έκθεση αυτή. Πριν ψηφίσουμε, και ελπίζω να μην φάμε πέντε ώρες αυτή την ψηφοφορία, με λίγη καλή τύχη. Θέλω να σας παρουσιάσω την ε, δήλωσή μας σχετικά με τον Brexit, που είναι ότι αποφασίσαμε στην έκθεση αυτή να μην αναφερθούμε στο Brexit. Και στην κοινή μας δήλωση θα σας εξηγήσουμε πώς περιμένουμε να συνεχίσουμε και ποια είναι η λογική μας για το Brexit. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι μετά την ψηφοφορία όλοι θα είμαστε λίγο χαρούμενοι, λίγο λιγότερο χαρούμενοι, αλλά όλοι θα στηρίξουμε την έκθεση αυτή για την φορολογία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λούντεκ, δίνω το λόγο στον συνεισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Λούντεκ και την ομάδα του. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις συζητητές, τη γραμματεία και τον Πρόεδρο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος ε, με την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο πλήρης έκθεση πάνω στο θέμα αυτό που έχει εκπονήσει ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβάλλει έτσι στις εργασίες του συνόλου της Επιτροπής με βάση όλα τα ευρήματά μας ε, κατά τη διάρκεια των αποστολών μας. Θα ήθελα να σας διαβάσω μία κοινή δήλωση των δύο συνεισηγητών, ε, του Λούντεκ Νίτερμαϊερ και δική μου, για το θέμα του Brexit, διότι είναι κάτι ε, για το οποίο έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες για την έκθεση. Θα σας διαβάσω λοιπόν την δήλωση την οποία θα λάβετε όλοι σας. Η ε, συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής, ε, πόσο μάλλον αυτού με του οποίου ασχολείται η Επιτροπή Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγή. Ε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η έκθεσή μας να υιοθετηθεί σήμερα από την Επιτροπή. Μέχρι το τέλος του Μαρτίου αλλά δεδομένης της πολυπλοκότητας της διαδικασίας του Brexit ε, έχουμε αποφασίσει να μην συμπεριλάβουμε συγκεκριμένη διατύπωση για το θέμα του Brexit αυτή τη χρονική στιγμή. Ο πρόεδρος διακόπτη. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ ακούστε αυτή τη σημαντική δήλωση. Αντιθέτως, ε, συμφωνήσαμε σε συντονισμό με όλες ε, τις πολιτικές ομάδες να ασχοληθούμε με το θέμα του Brexit ανάλογα με τη διαδικασία του άρθρου 50 της συνθήκης στο τέλος ε, του Μαρτίου, στην Ολομέλεια δηλαδή, ε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τότε. Η διατύπωση αυτή θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευση ανάμεσα στους συνεισηγητές και στους κοιόδες συνεισηγητές. Οι συνεισηγητές ε, χαιρετίζουν την εργασία που έχει γίνει από τις ομάδες διαπραγμάτευσης πάνω στα θέματα φορολογίας και Εφόσον συνεχίζεται η συζήτηση για τη φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπως δείχνουν οι γενικές συζητήσεις, όπως επίσης επιβεβαιώνουν οι διαπραγματεύσεις αυτής της ε, έκθεσης, υπάρχει ε, αυξανόμενη σύγκληση για πιο αποτελεσματική φορολογία, λαμβάνοντας υπόψη τις, ε, τις ε, συστημικές αλλαγές ε, στις οικονομίες και αυτό θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα φορολογικά καθεστώτα. Πιστεύω ότι μια τέτοια συζήτηση θα ξεκινήσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο εάν προχωρήσουμε στο Brexit και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάχει στη συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο ως μέλος της ΩΣΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και όλους για την καλή συνεργασία. Ο κύριος ε, ε, κύριε Πρόεδρε, ξέχασα να ευχαριστήσω και εσάς, ε, αλλά εάν καταφέρετε να ολοκληρώσετε την ψηφοφορία σε λιγότερο από πέντε ώρες, ε, θα σας ευχαριστήσουμε ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ωραία λοιπόν. Έχουμε τις εξής αντικαταστάσεις στο ΕΛΚ. Ριμπέιρο Σοφία αντικαθιστά τον Φερνάνδο Μανουέλ. Ε, επίσης, έχουμε την ε, Νίνα Τζίλ, Αγγιλέρα Κλάρα. που αντικαθιστά την Ανακομές. Ε, η Κλάρα Αγγιλέρα θα αντικαταστήσει την Ανακομέ. Ε, σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για ονόματα άλλων ε, αναπληρωτών ε, πριν ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Πιστεύω ότι όλοι έχουν τις κάρτες ψηφοφορίας. Αυτό ισχύει για όσους δεν είναι μέλη ή αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής μας. Σημειώνουμε όμως ε, την παρατήρησή σας. Απαρτία έχουμε ε, με το ελάχιστο 12 μέλη. Έχουμε απαρτία λοιπόν. Ας προχωρήσουμε σε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, να προχωρήσουμε στην δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Yeah, yeah, yeah, So what does it say? Is it fine? The vote is closed. Πέρα στις ψηφοφορίες. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1 και 1α. Ποιος είναι υπέρ? κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3, 3α, 3β, 3γ και 3δ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3E, 3F, 3G και 3H με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Έχουμε δύο παραπάνω από το ΕΛΚ, έναν παραπάνω από το ΕΛΚ από ό,τι θα έπρεπε. Ακυρώνεται η ψηφοφορία. Και θα ελέγξουμε τον αριθμό των μελών. Επαναλαμβάνουμε. Αρχή της ψηφοφορίας ε, για τη συμβαστική 3E, 3F, 3G και 3H. Αρχή της ψηφοφορίας, ονομαστική ψηφοφορία. λήξη της ψηφοφορίας. It's adopted. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3i και 3j. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61 με ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Έχουμε έναν ευρωβουλευτή παραπάνω από το ΕΛΚ, από ό,τι θα έπρεπε. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4, 4α και 4β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7α, 8 και 8α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές Συγγνώμη, διορθώνει ο Πρόεδρος. Συμβαστική 13 με ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. is open. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 και 15α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παρακαλώ μόλι. Ναι, θα με ακούσετε. Θα θέλαμε ονομαστικές ψηφοφορίες για τις τροπολογίες μας. Χρειαζόμαστε επαρκή στήριξη. Νομίζω την έχουμε, αλλά νομίζω ότι εννέα χρειάζονται για να έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Εάν θα μπορούσαν, σας παρακαλώ, οι συνάδελφοι να ψηφίσουν. Ε, μιλώ για την 15, αλλά το ίδιο θα ζητήσουμε και για όλες τις επόμενες. Τροπολογία 15. Θέλουμε ονομαστική ψηφοφορία. Παράγραφο 15. Τροπολογία 156, διορθώνει ομιλήτρια. Αναφέρεστε λοιπόν στην τροπολογία 156. Ποιος είναι υπέρ ονομαστικής ψηφοφορίας. Εννέα ψήφοι χρειάζονται. Ωραία. Πληρούνται αυτή η προϋπόθεση. Τροπολογία 156, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 175 υπέρ I'm afraid this one was not requested. Δεν έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία για αυτήν την τροπολογία πριν από την προθεσμία χθε. Ε, θα ψηφίσουμε λοιπόν για να τα σε 175 υπέρ, κατά, αποχές, η ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχή της ψηφοφορίας για την 175. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 και 17α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 20 και 20α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 και 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 230 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 241 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 με ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27, 27α και 27β. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28 και 28α. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Η λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 248. Μπορούμε να την ψηφίσουμε μαζί με την 251. Ωραία. Ψηφίζουμε τις δύο αυτές μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική 29. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 252 με ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 272. 273 και 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 33, 33α, 33β, 33γ και 33δ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 290 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 290 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 290 ψηφίζουμε. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 34, 34α, 34β και 34γ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 35, 35α, 35β και 35γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μόλι, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, Πίτερ. Και πάλι θα θέλαμε να ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία. Για να γλιτώσουμε χρόνο, προτείνω ε, να ρωτήσουμε τους συναδέρφους εάν συμφωνούν να γίνει ονομαστική ψηφοφορία για όλες μας τις τροπολογίες, διότι έχουμε άλλες εννέα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, 315 και οι άλλες τροπολογίες που ζητήθηκε από τους πράσινους να γίνουν με ονομαστική ψηφοφορία πριν την χθεσινή ε, προθεσμία. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν, έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Έχουμε νέα ψήφους. Ναι. 315 με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 36, 36α και 36β. Ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 326, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 36 γάμα, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Αρχή της ψηφοφορίας λοιπόν. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία. Μάλλον ηλεκτρονική επαλήθευση για την 176. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη. 1115 ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. So Uh, yeah, I'm afraid that it was rejected Απορρίπτεται. Uh, amendment 214. 214 ονομαστική ψηφοφορία. Oh, sorry. 218 roll call vote. The vote is open. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. And it was rejected. Απορρίπτεται. 214 ε, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 339 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 339, αρχή της ψηφοφορίας. How do we vote? The vote is closed. It's rejected. Λήξη της ψηφοφορίας. And it's rejected. Amendment 304. Απορρίφεται 342 και 343. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 727 ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος των πρασίνων. Yeah, in, in, in, in three parts. First part. Uh, first part. Until two. Okay. No? No? So what? Yeah, yeah. Yeah. Request to have the first part until DAC 2. Yeah. The, now we will vote on the first. Το πρώτο τμήμα μέχρι DAC 2. Ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται διότι γίνεται ψηφοφορία κατά τμήματα. Έχουμε ισοπαλία, αλλά είναι ψηφοφορία κατά τμήματα, δηλαδή σύμφωνα με τον κανονισμό εγκρίνεται. Η γραμματεία θα σας διαβάσει το σχετικό σημείο από τον κανονισμό. Ένα λεπτό θα το λύσουμε το θέμα. please, Under, under rule 117... Άρθρο 79α του κανονισμού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε κατατμήματα ψηφοφορία, σύμφωνα με το 176, θεωρείται ότι εγκρίνεται ε, το κείμενο. so second part. Yeah. Okay. So it's been adopted. Please quiet. Εγκρίθηκε λοιπόν. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ ησυχία. Μαθαίνουμε σιγά σιγά. Τροπολογία 727, ε, ε, το δεύτερο τμήμα μέχρι directive, ονομαστική ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. The third part by roll call vote. Τρίτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 348 υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Η ηλεκτρονική επαλήθευση 348. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, δεν είχαμε ισοψηφία. Συμβαστική 39 και 39α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 40, 40α, 41 και 42. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44, 44α έως 44i. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 379 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση. 379 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 798. Υπέρ, κατά, αποχές, η ηλεκτρονική επαλήθευση. 798, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 45, 45A και 45B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 407 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση. 407 αρχή της ψηφοφορίας. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 408 ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματο των πρασίνων. Αρχή της ψηφοφορία. ονομαστική ψηφοφορία για την 408. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 410 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 411 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 47 υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 413 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 419 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. έχει αποσυρθεί το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία για την 419 και ήταν πανομοιότυπη με την 420. 400, ε, συγγνώμη, συμβαστική 49, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 425, τροπολογία 425, υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. 425, αρχή της ψηφοφορίας, ηλεκτρονικός έλεγχος. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 426 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 435 από την τροπολογία 435 Για την 436 έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα την 435 για να ο σχηρός Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 436 με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε μαζί την 438, 439 και 440 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 52, 52A, 52B, 52C, 53 και ο τίτλος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 491 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση. 491, αρχή της ψηφοφορίας, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 54, 55 και 56 με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Συμβαστική 57, 58, 59, 59α και 59β υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 488 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση. 488 η ηλεκτρονική επαλήθευση αρχής ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Συμβαστική 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 575 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 64 και 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 520 Μάλλον όχι λέει ο πρόεδρος. Συμβαστική 68 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 528 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 529 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 70α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 70β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 537 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 71 και 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 74, 75 και 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 563 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 564 και 565 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. 564 και 565. Αρχή της ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 78α και 78β. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 80. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 584 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 595 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 667. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 86 και 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 87α. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 88. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 89. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 650. Η επόμενη είναι ονομαστική, οπότε δεν μπορούμε μαζί. Πρώτα την 650. Ε, το ισχυρό υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 653. Με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίπτεται. Και τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί 652, 651 και 654. Υπέρ, Καρτά. αποχές, απορρίπτονται. Συμβιβαστική 91 και 91α. Υπέρ, α, συγγνώμη, ονομαστική ψηφοφορία έχουμε εδώ, οπότε μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 91B με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 92 διανατάσεις ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 675 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 675. Ψεφίστε, παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Είναι γλωσσική η επόμενη. Συμβαστική 96 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 693. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 696 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 698 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 709 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ηλεκτρονικός έλεγχος 709. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 710. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 715 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 715. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 104 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 722 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 723. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 106. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 107. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 107α. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 108 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 744 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 110 και 110α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 748 με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 112, 112α και 112β. Υπέρ. Α, είναι ονομαστική ψηφοφορία αυτή. Οπότε ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 448. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. «758 τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Το έχουν ζητήσει οι πράσινοι. Μπορείτε να ψηφίσετε. 758. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 760. Υπέρ. Κατά. 760, ναι. Στην παράγραφο 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 112. C, D και ε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 767. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 766. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 768. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 769 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 770 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 773 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 115 και 116 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 778 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 779. Κατά τμήματα. Έχει ζητήσει το ECR. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα που αρχίζει με regrets και τελειώνει με finsen. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα is concerned αρχίζει μέχρι by the US one. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 116α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1194. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 777. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβαστική 116B. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 789. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 790. Υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 790. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 792. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 119 και 120. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 122. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 124 και 124α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβιβαστική 125 και 125α, νομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 826 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 126 και 126α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 127α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 843. Υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 128 και 128α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 129 και 129α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 129β και 129 γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 133α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 884 Οι συγγητές λένε για ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες, αλλά υπάρχει ονομαστική στο μεταξύ. Λοιπόν, 884 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 885 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 888 Ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 136α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 890 με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 891. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική τίτλος 5-5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 138, 138α, 138β και 138γ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβιβαστική 139 και 139α. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 141 και 141α υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 929 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 934 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 144 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 145 και 145α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 937 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 145β και συμβαστική 145γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 146 και 146α υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 862 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 943 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 944 τώρα και 945 γιατί είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για αυτές τις δύο τροπολογίες. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκαν. Συμβαστική 148 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 149 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 150 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 969 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 152 με ονομαστική ψηφοφορία μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 979. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβι... 980 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται να ελέγξουμε. Ωραία, θα ελέγξουμε για την 980 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 153. Υπέρ, κατά, αποχές. Έγκρινεται. Τροπολογία 973. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 154α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 992. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 998. Ονομαστική ψηφοφορία έχουν ζητήσει πράσινη. 998. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 1003. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 154D, δέλτα, με ονομαστική ψηφοφορία, μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 134 αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τις επόμενες τροπολογίες μέχρι την 138. Οπότε, ποιος είναι υπέρ των τροπολογιών αυτών. Κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Τέλος. Απορρίφθηκαν. Συμβαστική 155 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 156 μονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 192 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε για την 192 ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. The Τέλος. και απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 160 και 160α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 161α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 164 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1064. 1064 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για την 1064. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 167α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1079 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 170α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1097 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για την 1097 ψηφίζουμε τέλος Word. απορρίφθηκε 1093 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 171 και 171α υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 1114 ε, με ονομαστική κλίση που ζήτησαν οι πράσινοι άρχεται. Ψηφίζουμε για την 1114. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε αυτή τη φορά. συμβαστική 172. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε άρχεται τέλος απορρίφθηκε συμβιβαστική 100 17 17-28 ε, ε, η τροπολογία 11-18 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 11-19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11-20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11-21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11.22 Α, η 11.22 έχει αποσυρθεί. Οπότε ψηφίζουμε για την 11.23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 11.23. Άρχεται. Τέλος εγκρίθηκε 11-24 Πέρ, κατά αποχές αγκρίνεται όχι, συγγνώμη θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά you are right. You are right. Μάλιστα έχετε δίκιο. Η 11, 24 έχει καταπέσει. Η 1125 έχει αποσυρθεί και ψηφίζουμε για την 1126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Compromise 177. Συμβαστική 177. 177α και β. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ε, τροπολογία 1137. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για την 1137 τέλος απορρίφθηκε 1141 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβιβαστική 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 1149 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε για την 1149. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 179α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 180, 180α και β υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 1167 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για την 1167. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 181. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 181α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 181β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1184 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για την 1184. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται <clears throat> συμβαστική 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 1198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1199 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1208 υπέρ κατά αποχές ε, πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω. Ανεβοκατέβαιναν διάφορα χέρια. Λοιπόν, 12.08 ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε. Ένας παραπανίσιος από το ΕΛΚΑ. Για ξαναδοκιμάστε. Εντάξει τώρα. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας λοιπόν για τη 12.08. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 12.09 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστικές 192, 192α, β και γ, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστικές 195, 196 και 196α υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 1229 Προ... υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1232 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Γιατί τη 1232. Τέλος πληροφορια εγκρίνεται. 12.33 με ονομαστική κλίση άρχεται. Τέλος. Και εγκρίθηκε. Συμβαστική 200, 201 και 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 1242. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 1243 μέχρι και 1245. Unblock. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται απορριπτονται. Οπότε ψηφίζουμε για τη 12, 46, 7, 8, 9, 12, 50, 51, 52 οι οποίες είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 12-53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1254 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 1254 Τέλος της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Τροπολογία 1255 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε επίσης 12.55 άρχεται. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 335. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Πάμε στη συμβαστική 205 και 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική 207 μονοματιστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική για τα εκτιμώντας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τοποποιήθηκε, ε, με ονομαστική κλίση. Άρχεται, ψηφίζουμε. I close the vote. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συνεισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και όλους σας ε, για την προσήλωσή σας στην εργασία μας. Επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες που συνεργάστηκαν με την Επιτροπή μας και τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Ε, στην Ολομέλεια θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια του Μαρτίου, τη δεύτερη, στα τέλη Μαρτίου. Να κάνω μόνο μία παρατήρηση. Την περασμένη εβδομάδα παρακολούθησα δημόσιες εκδηλώσεις για το ξέπλυμα χρήματος και με εξέπληξε πώς εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των εθνικών κυβερνήσεων, δημοσιογράφοι, γνωρίζουν τις εργασίες της Επιτροπής μας, γνωρίζουν τις ακροάσεις που κάνουμε και επιπλέον και λένε πως ό,τι κάνουμε ε, ε, σημαίνει τη την εργασιες Είμαι πολύ περήφανος ε, που συνεργάζομαι με τόσο προσιλωμένους, αφοσιωμένους ε, συναδέλφους, γνώστες ε, των θεμάτων αυτών. Υπάρχει τίποτα στα διάφορα? Από ό,τι φαίνεται όχι. Να ζητήσω τότε από τους συνεισηγητές, εάν θέλουν κάτι να πούν, στο τέλος, όχι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στα διάφορα της Επιτροπής μας, οπότε πέρα στη συνεδρίαση σας ευχαριστώ πάρα πολύ.